Συνεχίζουμε τις επεξηγήσεις ψήφων. Επεξήγηση όσον αφορά την προγραμμάτισα των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ευρωεκφελιστικές ασθένειες. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Χουντής για ένα λεπτό. Δεν νομίζω ότι είναι παρόν ο κύριος Χουντής. Προχωράμε. Τώρα όσον αφορά την έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, Ζήτησε το λόγο ο, κυρία Μόρμπα η Κριστίνα. Είναι παρούσα. Θα ήθελα να μιλήσω ουγγρικά. Η έκθεση όσον αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες που είχα εγώ στην Ουγγαρία σαν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μιλάει για τα γεγονότα του φθινοπόρου του 2006 όταν η Ουγγρική αστυνομία ε, πετέθη κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σιωπηλή και παραμένει σιωπηλή η Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονό ότι η αστυνομία εξακολουθεί να, να, να συλλαμβάνει αυτού του ανθρώπου, να ενοχλεί αυτού του ανθρώπου ε, παράνομα. Και αυτή η παθητική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε σε αυτή την κατάσταση όπου 13 ε, μέλη της ε, αυτονών των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν συλληφθεί και παραμένουν σύλληψη διότι προσπάθησαν να ε, αποκαλύψουν περιπτώσεις διαφθοράς που διαπράττει η ισχύουσα κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση. Και τελικά καταπατεί η κυβέρνηση ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα των, ε, της αντιπολίτευσης. Έγιναν παράνομες έρευνες, οι υπολογιστές κατασχέστηκαν, χωρίς να τηρούνται οι νόμοι Και αυτά τα επανειλημμένως συνέβησαν χωρίς να αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καταψήφισα την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Στα πρακτικά της Τα πρακτικά θα υποβληθούν προσέγγιση του Κοινοβουλίου αρχές της επόμενης συνόδου. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, ήδη θα αποστείλω τα ψήφισμα, τα, θα καταχωρηθούν. Διακόπτεται η σύνοδος και καλό τέλος εβδομάδος σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.